εγκρίνεται η κυριότητα αυτών των εντολών. Ο κύριος Ρότζερ Χέλμερ μου είπε πως δεν είναι πλέον μέλος της ομάδας ECR και από 5 Μαρτίου ανήκει στην ομάδα Ευρώπη για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. Από το ΕΛΚ, τους Σοσιαλδημοκράτες, τους Φιλελεύθερους, το ECR και την QNGL μου ζητήθηκε να εγκρίνουμε τους ορισμούς ε, των ε, Προέδρων των Επιτροπών και Αντιπροσωπιών. Βρίσκονται οι ορισμοί αυτοί στα πρακτικά. Αν μέχρι τώρα συνεδρίαση δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, θεωρώ πως έχουμε εγκρίνει αυτούς τους ορισμούς. Σύμφωνα με το άρθρο